Colleagues, may I ask Συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε. Παρακαλώ συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Colleagues, we need to start Συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτή την πρώτη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Προπολογισμών για το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. είναι άκρος σημαντική στιγμή για αυτό το κοινοβούλιο, για αυτήν την θητεία και για τις επιτροπές μας. Το κοινοβούλιο μας ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευθετήσει το χάσμα επενδύσεων, να καλύψει το χάσμα επενδύσεων που είναι ένα από τα μείζωνα προβλήματα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οπότε καλωσορίζουμε την υποβολή πρότασης κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το γεγονός ότι η Επιτροπή αποφάσισε να ε, τοποθετήσει το πρόγραμμα επενδύσεων στο κέντρο των προτεραιοτήτων της. Καλωσορίζουμε επίσης το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε την κοινοτική μέθοδο. Έχουμε λοιπόν κανονισμό με την διαδικασία της συναπόφασης και γνωρίζουμε πλήρως τι διαδικασίες μας αναλογούν. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία και ο κανονισμός αυτός να ισχύσει ως το δυνατόν σύντομότερα προκειμένου το επενδυτικό πρόγραμμα Juncker να αρχίσει να λειτουργεί και να μπορέσει να στηρίξει την ανακάμπτουσα οικονομία. Ταυτόχρονα συνειδητοποιούμε τις ευθύνες μας και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορέσει να πετύχει αυτό το πρόγραμμα. Θα κοιτάξουμε να το βελτιώσουμε, να εξασφαλίσουμε το απαραίτητο επίπεδο δημοκρατικής ε, παρακολούθησης και ελέγχου και βάσει της εντολής που υπάρχει θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πετύχει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ώστε να δημιουργηθεί ταμείο με περιουσιακό με ενεργητικά στοιχεία που να βασίζονται στην εγγύηση των πόρων του προπολογισμού. Άρα το ε, Κοινοβούλιο έχει ιδιαίτερες ευθύνες εδώ. Είναι μια από τις δημοσιονομικές αρχές της Ένωσης, το σώμα μας. Όπως θα ξέρετε, ε, η διάσκεψη των Προεδρών αποφάσισε να ε, αναθέσει στις μεικτές αρμοδιότητες των Επιτροπών Οίκων και μπούτζ το θέμα αυτό. Οι επιτροπέ Ιτρέτα και Τραν συμμετέχουν βάσει του άρθρου 54 και επίση και άλλε ενδιαφερόμενε επιτροπέ θα ε, γνωμοδοτήσουν. Και συμμετέχουν βάσει του άρθρου 53 συν, όπως λέμε στη δική μας ιδιόλεκτο. Ε, έχουμε ήδη εδώ τους εισηγητές μας που θα κάνουν τις παρουσιάσεις τους, αλλά πρώτα-πρώτα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής Προπολογισμών, στον κύριο... Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που μπορούμε να συνεδριάσουμε εδώ οι δύο επιτροπές μαζί και μάλιστα θα έχουμε μαζί μας και την Τραν και την Ήτρε και άλλες επιτροπές. Και με τον τρόπο αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να καταδείξουμε ότι το Κοινοβούλιο είναι δυνατό όταν συγκλίνουν στις προτάσεις τους οι κοινοβουλευτικές επιτροπές αλλά και στις θέσεις τους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταδείξουμε, να αποδείξουμε ότι έχουμε την ικανότητα να πάρουμε γοργά αποφάσεις ε, οι οποίες ε, θα υποβοληθούν ε, στην Κομισιόν και μπορούμε γρήγορα να προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το νομικό εργαλείο το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στις επενδύσεις να ανθίσουν στο σύνολο της ενωσιακής επικρατείας και με τον τρόπο αυτό να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και στην ανάκαμψη της ανεργίας. Είμαι βέβαιος ότι θα εργαστούμε όλοι μαζί ε, και ε, με αμοιβαία επιφολή τρόπο. Και βεβαίως ξαναδίνω τον λόγο στον πρόεδρο Ρομπέρτο Γουελπιέρη Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε και μπορώ να ξεκινήσω με τον Ούντο Μπούλμαν από την ΕΚΟΝ. Vorsitzende, Αγαπητοί κύριοι πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμο κύριε συνάδελφο Φερνάντες, συν εισηγητή μου, αγαπητοί σκιώδεις εισηγητέ, σε Όλε τι αρμόδιε επίτροπε, Πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα που έχουμε αναλάβει σήμερα με την πρώτη κοινή μα συνεδρίαση. Όμως Πραγματικά πιστεύω πως και η απήχηση είναι εξίσου μεγάλη. Πολύ σωστά αναφέρατε πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωζώνη ακόμα δεν έχει φτάσει τα επίπεδα που είχε πριν την οικονομική κρίση όσον αφορά την οικονομική απόδοση. Έχουμε ένα τεράστιο επενδυτικό χάσμα στα κράτη-μέλη και στα δημόσια οικονομικά και στον ιδιωτικό τομέα. Και πραγματικά είχε φτάσει η ώρα να γίνει κάτι. Η πρωτοβουλία Juncker είναι κάτι που οφείλουμε να χειροκροτήσουμε και πιστεύω πως ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση συμφωνούμε όλοι γι' αυτό. Από όσο έχω συζητήσει μέχρι τώρα με τους κοιόδες εισηγητές. Όλοι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια καλή αρχή το συντομότερο δυνατόν. Φυσικά δεν πρέπει αυτό να θεωρήσουμε ότι σημαίνει πως υπονομεύεται η νομοθετική υπόσταση και η ποιότητα της δουλειάς μας, το ότι θέλουμε να δουλέψουμε γρήγορα δεν σημαίνει ότι δεν θα δουλέψουμε και καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποσαφηνίσουμε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια κατάλληλη λύση η οποία είναι απαραίτητη. Επιτρέψτε μου τώρα να κατονομάσω ορισμένα από αυτά τα πολύ σημαντικά προβλήματα στα οποία θέλουμε να βρεθεί μια λύση. Είμαι σίγουρος βέβαια ότι και ο συνάδελφος κύριος Φερνάντες και οι υπόλοιποι σκιώδεις εισηγητές θα λάβουν το λόγο και θα αναφερθούν και αυτοί σε αυτά. Φυσικά πιστεύω πως αυτό το ταμείο είναι ε, κάτι που έχει ανάγκη από ισχυρή χρηματοδότηση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό στην αρχή τουλάχιστον να υπάρχουν δύο πυλώνες, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από τη μία και ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη. Είναι φυσικά καλύτερο να υπήρχε μία ευρύτερη βάση, όμως οι συνάδελφοι της Επιτροπής Προϋπολογισμού θα ξέρουν καλύτερα από μένα τις λεπτομέρειες του σχεδίου αυτού χρηματοδότησης και τις εναλλακτικέ που υπάρχουν. Και αναφέρομαι στην Επιτροπή Μεταφορών, στην Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας. Γνωρίζω βέβαια και ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμού αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό ως πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, με πολλά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης. έργο δικό μας είναι να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το εξή ερώτημα. Τι γίνεται με την ποιότητα αυτής της πρωτοβουλίας, τι γίνεται με την ποιότητα αυτών των ε, νέων στρατηγικών, των νέων ε, επενδυτικών προϊόντων και σε τι διαφέρουν από αυτά που είδαμε μέχρι τώρα και από αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα. Τι λοιπόν είναι αυτό που χαρακτηρίζει ποιοτικά αυτή τη νέα επενδυτική στρατηγική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούμε για την ε, αντιμετώπιση, αντιμετώπιση μεγαλύτερων κινδύνων και αυτό φυσικά είναι μια πολύ συνετή προσέγγιση. Αλλά εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να ρωτήσουμε πώς θα το μετρήσετε αυτό και πώς μπορούμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνοδεύσουμε αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισης μεγαλύτερου κινδύνου. Και πώς θα αξιολογηθούν αυτά. Υπάρχουν κάποια συγκριτική αξιολόγηση, υπάρχουν άλλοι τρόποι έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε κάποια προϊόντα ως ιδιαίτερα επικίνδυνα και όχι ως ε, απλά συνηθισμένου κινδύνου. Έτσι ώστε να ενισχύσουμε την οικονομία. Είναι το μοναδικό κριτήριο το πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος ή υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Υπάρχουν ορισμένα ε, δύσκολα σημεία, υποδομές για παράδειγμα, ενεργειακή απόδοση. Υπάρχουν ερωτήματα τα οποία αφορούν πάρα πολλούς χώρους, τις υποδομές, τις μεταφορές. Υπάρχουν τομείς όπως αυτοί οι οποίοι χρειάζονται επενδύσεις και είναι και μάλιστα οι τομείς αυτοί οι οποίοι θα λειτουργήσουν όσο σκελετός έτσι ώστε να λάβει σάρκα και οστά, να λάβουν σάρκα και οστά αυτές οι επενδύσεις. Έπειτα, τα μέσα τα οποία έχουν προταθεί είναι τα κατάλληλα, έχουν τις κατάλληλες αρμοδιότητες έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι τους οποίους συζητούμε εδώ. Και εάν όχι, τότε θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Επίσης, θα πρέπει να δούμε όλες οι αρμόδιες επιτροπές, το πού βρισκόμαστε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτήν τη νέα θεσμική δομή που έχουμε μπροστά μας. Προβλέπεται μια στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πού στέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην διάθεση πόρων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Έχω ακούσει ότι, από κάποιους ότι ναι, είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε πόρους, όμως από την άλλη θέλουμε και μια εγγύηση ότι οι πόροι που θα διατεθούν θα επενδυθούν έξυπνα. Άρα δηλαδή τι θέλουμε, θέλουμε ίσα δικαιώματα στην απόφαση του πού θα δοθούν τα κονδύλια του προϋπολογισμού και σε τι επίπεδο, σε εθνικό, σε περιφερειακό, σε ευρωπαϊκό και ποια θα είναι η εμβέλεια του δικαιώματος συναποφασής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσοχή, αυτό που εννοώ είναι το ποιος είναι ο ρόλος μας ως εκπρόσωποι των λαών της Ευρώπης. Είναι λοιπόν έργο μας να προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε αυτές τις λεπτομέρειες και να εκπροσωπήσουμε τους πολίτες μας και για μένα είναι ξεκάθαρο ότι πραγματικά χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα από μία έκθεση μία φορά το χρόνο. Δεν μας φτάνει μία ετήσια έκθεση σχετικά με τον προϋπολογισμό. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες ενέργειες. Και τέλος. Πρέπει να πασχίσουμε να φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όλους τους ενδιαφερόμενους και να τους καθοδηγήσουμε στην έβρεση μια σωστή λύσης. Όμως η εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να διέπεται από μια καλή μίξη της πολιτικής πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε ανταγωνιστικές αγορές οι οποίες τώρα δεν είναι ανταγωνιστικές. Πρέπει να φροντίσουμε για σωστές υποδομές σε τομείς ιδιαίτερα όπου έχουν να κάνουν με συλλογικά αγαθά και πρέπει επίσης να έχουμε τη δυνατότητα να προβλέψουμε το ρόλο που θα παίξουν τα δημόσια οικονομικά σε τομείς όπου αυτή τη στιγμή δεν έχουν ανταγωνιστικότητα. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ώστε αυτή η ανταγωνιστικότητα να δημιουργηθεί για την αυριανή ημέρα. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρισκόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερα σημαντική θέση. Και δεν εννοώ μόνο ως ε, μέσω ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τους επενδυτέ, αλλά και ως διαμεσολαβητής έτσι ώστε να προσελκυθούν ιδιωτικές επενδύσεις. Thank you to... Ευχαριστούμε πολύ τον Ούντο Μπούλμαν. Τώρα θα δώσω το λόγο στον ε, συνεισηγητή από την πλευρά της ε, Επιτροπής, ε, τον κύριο Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, απλώς ήθελα να χαιρετήσω τους δύο Πρόεδρους των ε, Επιτροπών, καθώς και όλους τους συναδέλφους. Προφανώς, ε, μια ιδιαίτερη μνήμα ε, για τον συνεισηγητή, τον κύριο Μπούλμαν. Είμαι βέβαιος ότι όχι απλώς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, σε συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους εισηγητές, αλλά θα βρεθούμε στο των προσδοκιών των πολιτών, των προσδοκιών που έχουν αναποθέσει. Το πρόγραμμα αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ευκαιρία που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε χρησιμοποιώντας ότι υπάρχει στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Εδώ γυρνάμε τη σελίδα που τόσο πολύ περιμένουν και οι πολίτες να γυρίσουμε. Με αυτές τις επενδύσεις για την ανάπτυξη, με τις επενδύσεις για την απασχόληση. Το πρόγραμμα αυτό σε κάθε περίπτωση είναι συνέπεια της υπόσχεσης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά επίσης ε, και του αιτήματο που είχε εκφράσει επανειλημμένο στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε να ε, εγγυηθούμε ε, ένα ποσό 8 δις ε, ευρώ από τον προπολογισμό και να φτάσουμε τα 315 ε, δις ευρώ. Μπορούμε επιτέλους να κινητοποιήσουμε τους πόρους που υπάρχουν ως προς το ιδιωτικό χρήμα, αλλά να αναλάβουμε και μια πρόκληση. Μια πρόκληση που ε, πρέπει να αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο ευθύ αμέσω, ένα βραχή χρονικό διάστημα, όπου θα προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε εντό τη προθεσμίας που προτείνεται και αυτό το νομοθετικό ντοσχέ να φτάσει σε αίσιο πέρας και να καταφέρουμε να έχουμε μια συζήτηση πολύ ε, συνοπτική ώστε να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία στα τέλη Ιουνίου. Είναι μια πρόκληση για όλους όσοι είναι οι ενδεχόμενοι δικαιούχοι ε, αυτοί που θα υποφεληθούν από το πρόγραμμα προφανώς. Ε, δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανένα κράτος μέλος Θέλουμε όλοι να συμμετάσχουν ισότιμα και έμφαση πρέπει να δοθεί στην ιδέα της πλατφόρμας. Πλατφόρμας για την ε, συγκέντρωση των ε, προτινόμενων έργων, ώστε εκεί να διαρθρωθούν και να υλοποιηθούν τα διάφορα έργα και είναι και μια πρόκληση για την έρευνα. Είναι μια πρόκληση για την καινοτομία όχι μόνο για το γεγονός ότι οι επενδύσεις θα μπορούσαν να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα, τα πορίσματα της έρευνας, αλλά η έρευνα με τη σειρά της να τονωθεί και να αξιοποιήσει το κονδύλια του προγράμματος αυτού. Ως προς τους στόχους, υπάρχει ένα ευρύ πλαίσιο, διότι και στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020 θέλουμε βιώσιμες, ευφυείς, ε, επενδύσεις και βεβαίως ανάπτυξη που να επιτρέπει τη συμμετοχή όλων. Εδώ θα έχουμε πολλές παράπλευρες θετικές συνέπειες. Ευθύς αμέσως την υπέρβαση νομικών φραγμών ώστε να υπάρχει ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και βεβαίως μια σημαντικότατη στήριξη για τις επιχειρήσεις με λιγότερους από 30.000 εργαζομένους, ιδιαιτέρως για τις μικρομεσαίες. Σημειώνω ότι ε, το γεγονός ότι υπάρχει ευρεία συνένεση στο Συμβούλιο για την κατεπίγουσα ανάγκη να προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό είναι ένα σημαντικό ε, θέμα. Ε, ένα σημαντικό σημείο. Συνήθως ε, το Κοινοβούλιο είναι παρά τους εσωτερικούς διαχωρισμούς το πιο ενωμένο από το Συμβούλιο. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μια θετική ε, κίνηση και από το Συμβούλιο, μια θετική ένδειξη. Έτσι αυτό μπορεί να επιτρέψει την επιτυχία όλου του προγράμματος. Και τα σημεία που πρέπει εδώ να επιλύσουμε και που έχει αναφέρει και ο συνάδελφος Μπούλμαν δεν θα πρέπει να αποτελέσουν ένα, μια τροχοπέδη. Τροχοπέδη ώστε ε, το πρόγραμμα αυτό του 315 δις ευρώ να λειτουργήσει εγκαίρως. Και είναι μια πρόκληση και για τα κράτη-μέλη. Ε, ήδη ανέφερα τις πλατφόρμες επενδύσεων που θα μπορούσαν να ε, φέρουν πολλές επιτυχίες, ιδίως για τις δομές, τις ενεργειακές υποδομές, την ψηφιακή μας, το ψηφιακό μας θεματολόγιο. Όλα αυτά μπορεί εδώ να βρουν χώρο να αναπτυχθούν. Και επιπλέον πρόκειται για ένα πρόγραμμα που σε σχέση με τα όσα ήδη υπάρχουν μπορεί να συνδυαστεί με διορθωτικές ανάγκες είναι υποκαταστήσει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ευκαιρία την οποία πρέπει να δράξουμε. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα αντιλαμβανόντουσαν σε καμία περίπτωση πόσο ο της Ένωσης μπορεί να λειτουργεί ως εγγύηση και να μην υπάρχει καμία κίνηση προς τις επενδύσεις. Τώρα ελπίζουμε ε, ε, ότι θα ε, οδηγηθούμε σε αισιοπέρα εγκρίνοντα σύντομα το πρόγραμμα αυτό. Βεβαίω έχουμε τη δυνατότητα εδώ να βελτιώσουμε τόσα προτείνονται και αυτό είναι υποχρέωσή μα. Αλλά έτσι ενισχύουμε και τη δική μα την δημοκρατική παρουσία εδώ ε, συμμετέχοντας ενεργά στο πρόγραμμα αυτό. Ας σκεφτούμε τα υπόλοιπα ταμεία που υπάρχουν. Ε, μια ευρεία συζήτηση που τώρα μπορεί να ε, έχει μια θετική πυρια και σε αυτά τα ταμεία που ήδη λειτουργούν. Θέλουμε αξιοπιστία. Και ε, για την αξιοπιστία αυτή πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Απαιτείται μια διαρκής παρακολούθηση. Η διαρκής και συστηματική ε, εξέταση των όσων προτείνονται από το Ευρωκοινοβούλιο που ίσως και με την επίσκεψη ε, των ηθινόντων εδώ να διευκολύνει τα πράγματα. Προφανώς κάποια ζητήματα πρέπει να απαντηθούν, όπως η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων για τις Επενδύσεις, γιατί έξι και όχι περισσότεροι ε, εάν αυτή η Επιτροπή θα κάνει μια προεπιλογή των έργων, ε, εάν το Ευρωπαϊκό Ταμείο θα έχει προσέγγιση αποδοχής ε, θετικής αποδοχής των συστάσεων της Επιτροπής για τις επενδύσεις ή όχι. Θα πρέπει να είναι μια διεπιστημονική επιτροπή ή όχι αυτή των εμπειρογνωμόνων. Όλα αυτά θα τεθούν την κατάλληλη στιγμή. Όμως θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αυτό ε, ενισχύει, προσθέτει, βελτιώνει το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να τεθεί ένα αμφιβόλο αυτό το πολιτέ ε, πλαίσιο. Απλώς πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και υπάρχουν και άλλα ανοιχτά ζητήματα, όπως οι γραμμές. Οι γραμμές που θα λειτουργήσουν ως οριοθέτηση και θα επιτρέψουν να προσφέρει και εγγύηση στο επενδυτικό πρόγραμμα. Ή άλλα ζητήματα, ε, όπως ε, στόχοι του προγράμματος, το κέρδος, η απόδοση, αυτά εφόσον τα εγκρίνουμε θα πρέπει να κατευθυνθούν προς τις δημοσιονομικές γραμμές που τόσο πολύ έχουν πληγεί ως τώρα για έργα ή προγράμματα που δεν έχουν μπορέσει να λάβουν σάρκα και οστά λόγω της έλλειψης εγγύσεων. Εδώ χρειαζόμαστε ε, μία ε, προσέγγιση που να μας επιτρέπει ε, να μην διαταράξουμε την ισορροπία του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Με τόσα ανοιχτά ζητήματα βεβαίως και παρά το σύντομο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι είμαστε στη φάση που πρέπει να απαντήσουμε στις αγωνίες των Ευρωπαίων πολιτών και που έχουν αποθέσει σε εμάς τις ελπίδες τους τις ελπίδες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανταποκριθεί στην ανάγκη δημιουργίας ανάπτυξης, απασχόλησης μέσω των επενδύσεων και ότι θα κερδιθεί το στίχημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι με την συνεργασία που ήδη έχω δει να διαμορφώνεται θα καταφέρουμε να έχουμε συμφωνία και μάλιστα θετική εντός της προτινόμενης προθεσμίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε, κύριο, ευχαριστούμε κύριε Φερνάντες Και τώρα να ξεκινήσουμε με του από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ο κύριος Ατμαρκάρα. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά πιστεύω πως πρέπει να σπάσουμε όλες ε, τι συνήθειε και όλες τις τελετουργίε που έχουμε συνηθίσει με αυτήν τη συγκεκριμένη έκθεση. Αυτή η έκθεση αφορά κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας αφήσει να σκεφτούμε πολιτικά, κομματικά. Πρέπει να βρούμε μια κοινή προσέγγιση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να κάνω μια έκκληση να απαρνηθούμε από τώρα όλες τις πολιτικές κατευθύνσεις ή τις θεσμικές Διαφορετικά πιστεύω πως κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μία τρόπον την εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ μας στην ανάλυση αυτού του θέματος και τελικά να μην καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό το Ταμείο προσπαθεί να κάνει το ακατόρθωτο. Προσπαθεί να κινητοποιήσει αυτό που μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε και χρειάζονται τα κατάλληλα μέσα γι' αυτό. Και θα ήθελα να πω ότι υπάρχει αυτό που ακούμε και υπάρχει και αυτό που γνωρίζουμε και πιστεύω πως πρέπει να, να υπάρχει ανεξαρτησία πολιτική, ανεξαρτησία και καμία πολιτική επιρροή. διότι διαφορετικά δεν θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις για να φτάσουμε σε αυτό το ποσό των 315 δισεκατομμυρίων. Και επίσης να πω πως πρέπει και όλοι εμείς και τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουμε το ότι τα κονδύλια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και θα επενδυθούν στο κάθε κράτος μέλος θα ε, ε, επιστραφούν και όλες και ότι είναι αναγκαία και ότι κάθε λεπτό είναι αναγκαίο. Έχω ακούσει πολλές φορές για αυτή την συσχέτιση των επενδύσεων. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές το ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες και πιστεύω πως ε, χρειάζεται αυτή η ανεξαρτησία. Από τη μία έχουμε τα, τους ίδιους πόρους, τους ιδιωτικούς επενδυτές ανεξάρτητα project, ανεξάρτητη ανάθεση έργων και μετά αυτό που είναι δικό μας έργο είναι πώς θα οργανωθούν και θα συνδυαστούν όλα αυτά. Και τι ευθύνη έχουμε ως εκπρόσωπο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και ως Επιτροπή Προϋπολογισμού. Αλλά και ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Ποια ευθύνη λοιπόν έχουμε και ποια ευθύνη θέλουμε να έχουμε. Και πώς θα δράσουμε. Έπειτα, ένας άλλος τομέας στον οποίο ήθελα να αναφερθώ είναι ότι το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων πρέπει να βοηθήσει την ε, στην ανάληψη των ε, κινδύνων όμως δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να χρηματοδοτήσει ε, project για τα οποία τα κράτη-μέλη δεν διαθέτουν πόρους. Πρέπει δηλαδή να φροντίσει για μια de facto αηφόρο ανάπτυξη που θα δώσουν τα διάφορα έργα που θα χρηματοδοτήσει. Επίσης, οι επενδυτικές δυνατότητες για την ιδιωτική οικονομία πρέπει να χαρακτηρίζονται από ε, earmarking και να μην υπάρχουν ε, περιορισμοί και εμπόδια. Και σίγουρα αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί πάρα πολύ. Η πρόσθετη δηλαδή χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη, η οποία όπως είπα είναι αναγκαία. Και το σε ποια πλατφόρμα θα γίνει αυτή η χρηματοδότηση και ποιες συνέπειες θα έχει αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση και ποιες ε, θα είναι οι συνέπειες ε, που θα έχει στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η δική μου πολιτική ομάδα και εγώ προσωπικά πιστεύουμε ότι αυτό το ερώτημα του πώς δηλαδή ε, σχετίζεται όλο αυτό με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και, η... και πιστεύουμε ότι η ευελιξία αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να καθυστερήσουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δηλαδή, εξυγένση δημοσιονομική ε, και επενδύσεις πρέπει να ε, προσέξουμε να μην εμποδίζει η μία την άλλη. Χρειάζεται λοιπόν για όλα αυτά ένας ανοιχτός διάλογος και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα να κάνουμε συμβιβασμούς και ανάμεσα στις επιτροπές και ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες. Και ελπίζω κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του θέματος αυτού να μην χρειαστεί να συζητάμε κάθε φορά εκ νέου και την πάρα μικρή λεπτομέρεια σε κάθε μία αρμόδια επιτροπή. Αλλά να αναγνωρίσουμε την σημασία που έχει το να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα. Και πρέπει να πω ότι έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν αρκετά ταμεία τα οποία έχουν τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις. Και υπάρχει επίσης η εμπειρογνωμοσύνη που θα βοηθήσει και εμάς στο έργο της, στο έργο μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κάρας στόχος μας πράγματι ήταν το Κοινοβούλιο να είναι ενωμένο στο νομοθετικό αυτό έργο. Γι' αυτό και θα συνταχθεί μία έκθεση και θα δουλέψουν από κοινού οι δύο επιτροπές. Και πάντα θα έχουμε κοινέ συζητήσεις και μόνο κοινέ συζητήσεις. Για να είμαστε ενωμένοι πρέπει να υπάρχει αυτοπιθαρχία στη χρήση του λόγου και βέβαια να συζητούν οι συνάδελφοι τον περισσότερο μεταξύ τους. Για σήμερα θα ορίσω ως χρόνο αγόρευση στα τρία λεπτά. Εκ μέρους της Δημοκρατικής Ομάδας από την Επιτροπή ΕΚΟΝ, η κυρία Ιντέρ. Γκόρθαρ είναι η εισηγήτρια αλλά αντικαθίσταται σήμερα από την Ιζαμπέλ Τομά. Ευχαριστώ πολύ κύριοι πρόεδροι. Φυσικά και μας ικανοποιεί η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σε σχέση με τον προτινόμενο μηχανισμό. Και τα προβλήματα αυτά πρέπει να επιλεφθούν τάχιστα. Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, καταρχάς να πω ότι η κυρία Γκουαρθιάμπα δεν είχε προβλέψει αυτή την αλλαγή ημερομηνία, γι' αυτό και δεν είναι εδώ ό,τι αφορά τον νοσιακό προπολογισμό δεν υπάρχει πρόβλημα σχετικά με το ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνετάσχει σε αυτό το επενδυτικό σχέδιο. Με τον τρόπο αυτό άλλωστε θα έχουμε και καλύτερη συναπόφαση, πράγμα που μας χαροποιεί. Ωστόσο αναρωτιόμαστε λίγο για τις επιλογές που έχουν γίνει ορίζοντας 2020 και μετά ε, το Connecting Europe. Αναρωτιόμαστε εάν και κατά πόσον είναι οι σωστές επιλογές. Δεν πιστεύουμε ότι θα είναι ανώδυνες αυτές ε, οι επιλογές για τα υφιστάμενα προγράμματα και επομένως είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό. Επίσης όσον αφορά τα 21 δις ε, το βασικό κεφάλαιο λοιπόν και εδώ αναρωτιόμαστε βρισκόμαστε ε, σχετικά με αυτό το βασικό κεφάλαιο και για το κατά πόσον δηλαδή αυτό ε, το κεφάλαιο είναι αρκετό. Ε, το Συμβούλιο είπε ότι δεν θα υπάρξει συμμετοχή των κρατών μελών και επομένως μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά αυτήν την επιλογή που έκανε το Συμβούλιο και επίσης αναρωτιόμαστε εάν και κατά πόσον θα πρέπει να βρεθούν τρόποι να διευρυνθεί αυτό το βασικό κεφάλαιο για τους λόγους που εξήγησα ήδη ε, και όσον αφορά και το, τον μοχλό, το, το αποτέλεσμα του μοχλού που θα πρέπει να έχει. Τώρα, συμφωνώ απολύτως με αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, ε, δηλαδή το θέμα των κρατών μελών δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόσκομα στην ε, επιλογή των πιο αποτελεσματικών και καλών προγραμμάτων ε, θα, είμαστε, θα επαγρυπνούμε ε, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη και τα προγράμματα τα οποία περισσότερο πρέπει να γίνουν ε, εκεί ακριβώς να προωθούνται οι, τα κονδύλια. Τέλος, αναρωτιόμαστε εάν υπάρχει πραγματικά καλή σχέση και αντιστοιχεία ανάμεσα ε, στη νομική βάση, το άρθρο 5 και ε, ε, το γενικότερο εγχείρημα. Η Κομισιόν αναφέρεται σε ένα νέο προφίλ κινδύνου που λαμβάνει υπόψη και την ενεργειακή μετάβαση, που λαμβάνει υπόψη τις θέσεις εργασίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εμείς ακόμα και την κατάρτιση που αναφέρεται στο 5 και αναρωτιόμαστε εάν αυτές οι αυτοί οι επενδυτικοί προσανατολισμοί ε, μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν μοχλό για να προχωρήσουμε καλά. Επίσης, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, και συγκεκριμένα όσον αφορά την προσθετικότητα αυτού του ε, ταμείου σε σχέση με τα ήδη υφιστάμενα ε, δεν είμαστε βέβαιοι ότι συμφωνούμε απολύτως με τον τρόπο με τον οποίο αυτό το ταμείο θα έρθει να προσθεθεί στα υφιστάμενα. Ε, πο, πολλοί είναι οι προβληματισμοί μας επίσης και όσον αφορά τους μακροοικονομικούς στόχους και θα πω μόνο το εξή πώς θα μπορέσουμε τις τοπικές και εθνικές επενδυτικές τράπεζες οι οποίες ε, βοηθούν περισσότερο πιο κοντά στις επιχειρήσει πώ πώς θα τις εντάξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Παίρνω τώρα το μικρόφωνο εγώ στη θέση του Προέδρου από τον Ρομπέρτο. Έχουμε ακόμα 13 παρεμβάσεις και στις 7 όμως θα πρέπει να σταματήσουμε. Ε, άρα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει δύο και ο καθένας έτσι ώστε να μπορούσαν να μιλήσουν όλοι. Σάντερ Λούνς. Ευχαριστώ πολύ. Θα κερδίσουμε χρόνο, θα μιλήσω Ολλανδικά. Ε, γιατί ούτως ή άλλως ε, λείπει η συνάδελφος που είναι ε, λειπει η που ειναι ε υπευθυνη για την δεύτερη επιτροπή. Θα μιλήσω μόνο εγώ θα μιλήσω βέβαια εξ ονόματός μου. Εμείς διαβάσαμε όλα τα έγγραφα τα οποία κυκλοφόρησαν στη διάρκεια της προηγούμενης συζήτησης και ό,τι κυκλοφόρησε και το Συμβούλιο. Εγώ θα ήθελα ε, να αναφερθώ σε συγκεκριμένα θέματα. Πρώτον, ε, είναι ορθό ότι ε, θα πρέπει να ε, κατανοούμε ότι η, λύση όλων των προβλημάτων αυτής της μηχανής της οικονομίας που δυσκολεύεται να πάρει μπροστά δεν είναι απλώς να ρίξουμε στη μηχανή αυτή χρήματα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν και διαφορετικέ μεταρρυθμίσει έτσι ώστε ή ταυτόχρονα και, μετα, και μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε ε, η οικονομία να πάρει μπροστά. Δεύτερον, ε, ποιον προπολογισμό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για αυτό το ταμείο ε, ε, Συνειδητοποιούμε ότι εδώ προσπαθούμε να δούμε τα χρήματα τα οποία έχουν επενδυθεί μέχρι τώρα στον ε, τομέα αυτό. Δεν μπορούμε να βρούμε χρήματα ας πούμε αλλού. Ε, διαπιστώνουμε ότι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά μήπως ε, και σε άλλα σημεία του προϋπολογισμού της Ένωσης μπορούμε να βρούμε και κάποια ε, χρήματα τα οποία να μπορούν καλύτερα να χρησιμοποιηθούν. Ε, γιατί αναφερόμαστε στον παράγοντα 15 ας πούμε. Τρίτον, αυτό το ταμείο θα πρέπει να είναι μόνιμος μηχανισμός ή πρόσκαιρος. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι πρόσκαιρος γιατί παρουσιάζει στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να είναι ε, μόνιμα αν θέλουμε να είναι πραγματικά αποτελεσματικά. Όταν ε, θα έχει επιτευχθεί ο στόχος θα πρέπει να σταματήσει ε, να υπάρχει αυτό το ταμείο όσον αφορά τα συγκεκριμένα προγράμματα. Να πω το το είπε το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη τα οποία συμβάλλουν ε, στην δεξαμενή έργων θα μπορούν να ε, έχουν μεγαλύτερο λόγο στην επιλογή των ε, έργων. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι σημαντικό. Ο κύριος Καμάλ έχει πει ότι οι αρχές δεν μπορούν να παίζουν σαν να είναι καζίνο και επομένως τα ε, θα πρέπει ε, να είμαστε σίγουροι ότι δεν ε, χάνει, αν, χαθούν τα χρήματα δεν θα τα χάσουν οι φορολογούμενοι. Κύριε Πρόεδρε. Eh λοιπόν, ο επόμενος ομιλητής δεν είναι εδώ. Ραμόν Τρεμόσα ή Μπαλσέλς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε λεπτό θα πω αυτά που θέλω να πω. Βεβαίω με την καλύτερη των διαθέσεων ε, ακούω αυτήν την ε, πρωτοβουλία που θα μπορέσει να δώσει στην Ευρώπη 300 ε, και πάνω δις και που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Σε πολλά κράτη-μέλη, κυρίως στην Νότια Ευρώπη, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε δει ε, μεγάλες ε, περικοπές ε, των ε, δημοσίων ε, δαπανών ε, και έχουμε μία στροφή αντί για αμυντικές δαπάνες ας πούμε έχουμε κάποιες επενδύσεις σε άλλους τομείς. Τώρα βέβαια ο τρόπος με τον οποίο κανείς επενδύει τα χρήματα που έχουν προκύψει από τις περικοπές αυτό είναι φιλοσοφικό ερώτημα ε, το σημαντικό ε, ερώτημα είναι πώς θα χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα αυτά. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να σταματήσουμε πια να επενδύουμε σε τρένα χωρίς επιβάτες, σε αεροδρόμια χωρίς αεροπλάνα και επομένως σε ανώφελα έργα γενικά θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτά τα έργα τα οποία έχουν έχουν ήδη ξεκινήσει τα τελευταία πέντε χρόνια. Ας πούμε στην Επιτροπή Μεταφορών έχουμε απομονώσει πολλά ε, σημαντικά έργα τα οποία ε, στον τομέα των μεταφορών έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία. Υπάρχουν κάποια project σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο οποίο ήδη τα τρία θεσμικά όργανα επενδύουν χρήματα με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει τουλάχιστον αυτά να προωθηθούν και να μην δώσουμε ρόλο και λόγο σε ορισμένες πρωτεύουσες να πάρουν αποφάσεις οι οποίες ενδεχομένως θα αντιτίθενται στο ευρωπαϊκό συμφέρον. Ε, Νίλ Τόβαλς. Ευχαριστώ πολύ. Έχω έξι σημεία. Το πρώτο είναι, είναι μόνιμη ή προσωρινή λύση αυτή. Όλοι λένε ότι είναι μια προσωρινή λύση, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι ο κόσμος ευρύθη προσωρινών λύσεων που είναι για 4, 40, 50 ή και 200 χρόνια μαζί μας τελικά. Άρα μάλλον μιλάμε και εδώ για κάτι μόνιμο. Έρχομαι στο δεύτερο σημείο. Εάν είναι ένα μόνιμο ταμείο, θα πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα εξεύρουμε τους σπόρους για αυτό το ταμείο. Και όχι μόνο να δούμε ποιο είναι ο πιο εύκολος τρόπος για την εξέβριση σπόρων για αυτό το ταμείο. Τρίτον, τίθεται ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα για το πώς αποδοτικά θα δαπανηθούν οι πόροι αυτοί. Και όταν στο μέλλον θα συζητήσουμε τον προπολογισμό θα πρέπει να δούμε τα χρήματα, θα τα δίνουμε έτσι τσάμπα ή ως ε, μια μορφή δανείου για να είναι πιο αποτελεσματική η διάθεση αυτών των χρημάτων. Το επόμενο. Τα χρήματα, τα κονδύλια των θεσμών. Αγωνιστήκαμε για αυτό το πολιτές μισονομικό πλαίσιο και ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν χρήματα. κάποια στιγμή βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα όμως τα κράτη-μέλη χρήματα, αλλά τα δικά μας χρήματα, όχι τα δικά τους. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα, το πόσο εύκολα βρίσκονται αυτά τα ε, χρήματα. Επόμενο, ήδη οι πόροι. Εάν δεν πετύχουμε αυτή τη φορά να καταλήξουμε στου ίδιου πόρου, δεν θα το πετύχουμε ποτέ. Πρέπει λοιπόν να ρυθμίσουμε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν στου ίδιου πόρου. Και τελευταίο, έκτο, Κάθε μέρα μιλάμε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά δεν κάνουμε και πολλά. Κάνουμε ελάχιστα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει τέλε, επαφή είπε ο Μπούλμαν. Πράγματι, αυτό χρειάστηκε στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και έμεινα στα δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριο. Μπα Χέικχαουτ. <clears throat> Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι υπάρχει φυσικά η επιθυμία των μεγάλων πολιτικών ομάδων για σταθερότητα και ρύθμιση, όπως για παράδειγμα με το, με το σύμφωνο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Πρέπει να δούμε και τις ε, υπόλοιπες ε, πτυχές και να σας πω ότι αυτά τα δύο λεπτά μου φαίνονται λίγα. Όπως και να έχει. Ε, πραγματικά θα χαρώ πολύ να συμμετέχω σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων μη ιδεολογικού χαρακτήρα. Και φυσικά συμφωνώ και εγώ ότι χρειάζονται επενδύσεις και ότι οι επενδύσεις χρειάζονται πολύ περισσότερο σε μέρη όπου έχουν πληγεί πολύ περισσότερο από τις ε, ε, πολιτικές λιτότητας και πρέπει να το τονίσουμε αυτό όταν θέλουμε να μιλήσουμε για επενδυτικά πακέτα. Έπειτα να χρειάζεται, αν, χρειάζεται να δούμε τι θα γίνει και με τα επιτόκια. η πρόταση Juncker μιλά για δημόσιες ε, και ιδιωτικές επενδύσεις, όμως αυτό κοστίζει πάρα πολύ στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Για παράδειγμα, φτιάχνεις έναν αυτοκινητόδρομο, ο οποίος δεν αποφέρει έσοδα και πώς θα τον κάνεις κερδοφόρο, θα βάλεις διόδια. Ε, όταν θέλεις να εξοικονομήσεις ενέργεια και χρειάζεσαι έναν ε, επενδυτή πρέπει ε, να, δούμε τι γίνεται με τα επιτόκια. Όταν είναι μηδενικά τα επιτόκια, λογικά δεν θα μπορέσει να προσελκύσει πιο δύσκολα επενδυτές. Φυσικά οι πολιτικές λιτότητας έχουν επηρεάσει διαφορετικά τον καθένα και πρέπει να δούμε πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι επενδύσεις με νέα δάνεια, με αυξημένη φορολόγηση των ε, μεγάλων ομίλων. Αυτά είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να μας ε, απασχολήσουν. Επίσης, επενδυτικά ομόλογα. Πρέπει να δούμε λοιπόν και αυτές τις, τις πτυχές. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μισό λεπτό, λέει ο κύριο Σέικχαουτ. Να επισημάνω, Πρόεδρε, ότι μίλησε η Γκουε και όχι ο κύριο Μπα Έκχαουτ, για να ξέρετε τι γίνεται και με τον κατάλογο των αγορητών. Συμφωνώ με τον Φάμπιο, αλλά έπρεπε να το πω. Δεν έχω σωστό τον κατάλογο, ίσω, ε, βάσει τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και τη σωστή σειρά. Γι' αυτό πήρε το λόγο όντω ο κύριο Δεμάζη. Ο κύριο Μαραγκάλ. Ευχαριστώ. Προεδρή. Για να δούμε. Μιλάμε για το πώς ιδιωτικά κονδύλια θα τα βάλουμε να υπηρετήσουν το ομοσπονδιακό συμφέρον. Αυτό είναι το σχέδιο. Πώς θα κινητοποιήσουμε ιδιωτικές επενδύσεις ε, για να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον. Ποτίθεται ότι είναι άφθονα και διαθέσιμα τα χρήματα αυτά, αλλά θα εμφανιστούν αυτοί οι πόροι μόνο αν έχουμε εγγύηση ή αν είναι αμοιβεοποιημένες οι απώλειες. Και βέβαια αυτό ε, απριόρι μας φαίνεται απαράδεκτο. Αλλά θέλουμε αυτό το ταμείο να μην είναι απλά ε, προσδοκίες και αν θέλουμε πραγματικά να αναθερμάνει την οικονομία θα πρέπει να το ενσωματώσουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο γενικής οικονομικής πολιτικής. Να αφήσουμε κατά μέρο τα δόγματα που ακόμη κυριαρχούν, απαρότι φαίνεται απόλυση, ενδείξει τουλάχιστον ότι δεν αποδίδουν. Μόνο αν το Ταμείο εξπετήσει κοινό στόχο θα μπορέσει να δημιουργήσει κατάλληλε προποθέσει ώστε κάθε κράτο μέλο να μπορέσει να ακολουθήσει το μονοπάτι το αναπτυξιακό εξόδου από τις κρίσεις και να δημιουργήσει και εκ νέου το ευρωπαϊκό παράδειγμα ανάπτυξης και ε, δημιουργικότητας. Υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες εγγύσεις. Πρέπει να ορίσουμε ε, το ποιος θα αποδίδει λογαριασμό, η λογοδοσία θα πρέπει να είναι συστηματική. Από πού θα προέρχονται αυτοί οι πόροι της αρχής εγγύησης, από ποια κονδύλια. Δεν συμφωνούμε με την αρχική πρόταση, το πρόγραμμα Horizon ή το 2020. Ποιες είναι οι βασικέ προποθέσει του σχεδίου, Κατ' εμάς Θα πρέπει δύο να είναι τα βασικά κριτήρια. Πραγματικές επενδύσεις, να έχουμε έναν λογικό κίνδυνο και έπειτα να επιδιώκονται κοινωνικοί στόχοι. Δηλαδή να δημιουργήσουμε βιώσιμες θέσεις εργασία παραδείγματο χάρη. Δεν μπορεί να περιλαμβάνονται στο σχέδιο οτιδήποτε θέτει σε κίνδυνο την παροχή των δημόσιων κοινοφελών υπηρεσιών. Ούτε πρέπει να υπάρξει ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Και αν υπάρχει θα πρέπει αυτά να είναι η ενέργεια, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Ο στόχο είναι να προωθήσουμε την εσωτερική ισορροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριο Μπά. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω κάτι στα ένα-δυο σχόλια που έγιναν. Ακούστε και από το ΕΛΚ ότι δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια ιδεολογική συζήτηση εδώ, θεωρητική, που ωραία είναι να την ακούει κανεί, γνωρίζοντα κιόλα ότι το ΕΛΚ ε, πάντοτε επέκρινε η επένδυση. Τώρα θα μπορούσε να ξεκινήσει και μας λέει ότι δεν θέλει μια ιδεολογική συζήτηση. Το ΕΛΚ ε, μιλά για πρόγραμμα ξένων επενδύσεων, θα το καλωσορίζαμε, αλλά πρέπει να δούμε και το ύψος φιλοδοξιών του προγράμματος. Ξέρω ότι η ΑΛΔΕ έχει προτείνει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 700 δις, ε, το, οι σοσιαλιστές 800. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο αυτή την πρόταση και να την κάνουμε φιλοδοξότερη. Καλωσορίζω την προσέγγιση του ΕΛΚ ότι δεν θα τοποθετηθούν ιδεολογικώς στην όλη κουβέντα. Πολύ καλό αυτό και όντως μακάρι να το κρατήσουν. Ε, τώρα για τα διάφορα σημεία του προγράμματος που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του επενδυτικού προγράμματος. Πραγματικά πρέπει να κάνουμε μια ε, συνολική συζήτηση για τον ε, παράγοντα μόχλευσης του 2015. Ε, στα χαρτιά έχουμε 315 δις, αλλά ξέρουμε ότι προ στιγμή έχουμε μόνο 21 δις στο πρόγραμμα. Από πού θα έρθει λοιπόν αυτός ο παράγοντα μόχλευση. Εκεί ικανό θα είναι να γίνει μια εντελεχή συζήτηση. Και επίση, εάν δούμε την επιλογή των έργων. Εκεί έχω σοβαρέ αμφιβολίε για την έλλειψη κριτηρίων. Για, την, ε, για το πώ ε, προσθέτουν μεταξύ του τα έργα, ποια είναι τα κριτήρια, ε, πώ το κίνδυνο ενδεχομένω τον, τον αναλαμβάνει το κοινό, ενώ ιδιωτικό τομέα μόνο το κέρδο. Και επίση, μήπω το Horizon 2020 και το, η διευκόλυνση για την διασύνδεση τη Ευρώπη αποστερούνται των ε, πόρων που του αναλογούσαν. Θέλουμε να είμαστε ενωμένοι, αλλά βεβαιωθούμε ότι το Κοινοβούλιο το, τελικά εγκρίνει ένα, πραγματικό καλό, ένα πραγματικά καλό πρόγραμμα που δίνει αποτελέσματα και α μείνουμε όντω μακριά από κάθε ιδεολογική συζήτηση. Χαίρομαι που θα ακολουθήσουν αυτή την ανιδεολογική συζήτηση μαζί μα ε, όλοι οι πρόσωποι του ΕΛΚ. Σα ευχαριστώ, κύριο Ζάνη, ο οποίο ε, θα είναι εισηγητή εξ τη Επιτροπή Προπολογισμών αλλά και εξ ονόματος της ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ίσως λοιπόν ε, ε, να έχω και λίγο περισσότερο χρόνο. Τα στοιχεία τα οποία ανέφεραν οι συνάδελφοι και τα σημεία τα οποία έδειξαν είναι πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ ε, ευνοϊκά δέχομαι αυτή την πρωτοβουλία, αλλά είμαι ιδιαίτερο επιφυλακτικός, διστακτικός όσον αφορά το καλό αποτέλεσμα που μπορεί να έχουν τέτοιου είδους προτεραιότητες. Εγώ θα έλεγα ότι παρά να δημιουργούμε τέτοιου είδους μηχανισμούς σε ενωσιακό επίπεδο ε, για να ενισχύσουμε τις επενδύσεις, ίσως καλύτερα θα ήταν να, δώσουμε, να αφήνουμε, να δίνουμε περισσότερο περιθώριο ελιγμών στον προπολογισμό των κρατών μελών έτσι ώστε να κάνουν τέτοιου είδους προγράμματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς από την Επιτροπή Προϋπολογισμών λέμε ότι θέλουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να δούμε τους ε, πόρους που θα βγουν ας πούμε από το, Horizon, από ε, ε, το πρόγραμμα Horizon 2020. Δεν θέλουμε τα προγράμματα από τα οποία ε, θα ληφθούν χρήματα να έχουν πρόβλημα τα προγράμματα αυτά. Δεν είναι δυνατόν προγράμματα τα οποία έχουν ήδη ορίσει ως προγράμματα προτεραιότητας και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και οι χώρες να μείνουν χωρίς χρήματα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν ότι προγράμματα τα οποία είναι πρωταρχική σημασίας ε, δεν θα ε, ε, αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Απ' την άλλη πλευρά 21 δις, αυτά είναι λίγα και σαν εγγύηση είναι λίγα. Δεν είναι δυνατόν εμείς να βασιστούμε σε ένα τόσο μικρό αρχικό ποσοστό γιατί από το 2011 και μετά ο ιδιωτικός τομέας δεν επενδύει και δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή οι ε, προϋποθέσεις έτσι ώστε να ξαναρχίσει να επενδύει ο ιδιωτικός τομέας. Διαφάνεια, απαραίτητη διαφάνεια και όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων αλλά ε, και στην ταυτοποίηση του ποιος συμμετέχει, ποιος ε, ε, θα συμμετάσχει από πλευράς ε, του δημόσιου, από πλευράς του ιδιωτικού τομέα. Αυτά τα ομόλογα έργου, τα project bonds, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ένα είδος μετακύλησης ευθύνης ε, των προγραμμάτων αυτών. Μας απασχολούν κυρίως εάν και πώς μπορούν να καλυφθούν αποτυχίες στην εκτέλεση των project αυτών. Επίσης ε, ε, η γραφειοκρατία, εάν θέλουμε, η διακυβέρνηση μάλλον, εάν θέλουμε να μην επιβαρυνθούν τα προγράμματα αυτά με μεγάλη γραφειοκρατία, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει πιο ευέλικτη η διακυβέρνηση. Και κάτι άλλο που θέλω να μου διαλευκάνετε, ε, τον αντίκτυπο στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ταμείου αυτού, επί του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα τρία χρόνια. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ναι, ε, είναι εισηγητή και από την ΕΚΟΝ και από την πούτσα, Επομένω, ε, του δίνουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Ε, έφτασα στο τέλο. Περαίνοντα λοιπόν να πω ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στους δύο από τους τρεις πυλώνες που αναφέρει η Κομισιόν. Ε, δηλαδή να στοχεύσουμε σε ε, προτεραιότητες ε, οι οποίες θα οδηγήσουν στην βιώσιμη ανάπτυξη. Μας αρέσει αυτός ο όρος. Δεύτερον και πιο σημαντικό θα πρέπει να δούμε το θέμα της άρσης των προσκομμάτων έτσι ώστε πραγματικά ο ιδιωτικός τομέας να επανεπενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Λιάννη Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μιλήσω το πολύ ένα δίλεπτο για να καλύψω την υπέρβαση των συναδέλφων. Θα ήθελα οι συνεισηγητές να σκεφτούν ότι εξαιτία της ταχείας διαδικασίας θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μπορέσει να λειτουργήσει η πρόταση αυτή, να πετύχουμε τις δύο Υπάρχουν πολλά σημεία που πρέπει να δούμε, όπως πολλά ζητήματα δεν μπορούμε να τα ορίσουμε ποσοτικώς. Θα πρέπει όμως να βεβαιωθούμε και για την δημοκρατική μας λογοδοσία, ιδίως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία ε, και ανάληψη ευθυνών, καθώς και διαφάνεια ε, και ε, σωστός καθορισμός των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας. Πώ θα έχει σωστή πρόσβαση στι πληροφορίε το κοινό όμω. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι χώρε που δεν θέλουν ιδιωτικού επενδυτέ. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια σωστή διαθέτηση και να βεβαιωθούμε ότι όλα τα κομμάτια του παζλ ταιριάζουν. Διότι οι στόχοι πρέπει να είναι ε, παρόμοιοι. Δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση πρόχειρη βάρο προγραμμάτων όπω το Horizon 2020 τη διευκόλυνση και την σύνδεση τη Ευρώπη. Και σε καμία περίπτωση να μην ξεχνάμε του φορολογουμένου που τελικώ αυτοί θα αναλάβουν το μεγαλύτερο βάρο. Ευχαριστούμε και τώρα να ακούσουμε τους εισηγητές των επιτροπών, των ε, συμμετοχουσών επιτροπών βάσει του άρθρου 54. Από την Ήτρε η κυρία Βαν Μπρέντ. Νομίζω ότι μόλις βγήκε από την αίθουσα όμως. Ο κύριος Ρικέ από την Επιτροπή Τραν έφυγε και εκείνος. Είναι εδώ. Α, ήταν, ήταν εδώ. Όμω η κυρία Ενέσα Γιάλα Σέντερ είναι εδώ. Έχετε το λόγο, κυρία Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να μην χάσω τελείω τη φωνή μου μέσα σε αυτό το λεπτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσετε τη δυνατότητα να μιλήσω σε αυτή τη συνάντηση των δύο αρμοδίων επί επιτροπών. Η Επιτροπή Μεταφορών ήδη συζήτησε σε βάθος το θέμα αυτό. Νομίζω ότι οι πολιτικές ομάδες λίγο πολύ είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Θέλουμε να σας εκφράσουμε την ανησυχία που έχουμε σε σχέση με την απόφαση ε, που μετά από τρία χρόνια ελήφθη και μετά από το διάλογο για αυτό το χρηματοπιστωτικό μέσο που ήδη έχουμε, το χρηματοδοτικό μέσο, το Connecting Europe Facility. 26 Φεβρουαρίου λίγη προθεσμία για τους πρώτους διαγωνισμούς ε, αξίας 6 δις για τις υποδομές δηλαδή που έχουν συμφωνήσει μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και με τις περιφέρειες ε, και άλλους ε, φορείς. Επομένως, για μας, με βάση την πρόταση της Κομισιόν, που δίνουμε το 1 τρίτο από τα 8 δις που προβλέπετε στο βασικό προϋπολογισμό στο Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Εμείς λοιπόν εκφράζουμε την ανησυχία μας σε σχέση με το τι πρόσθετο όφελος ή ποια είναι η διαφορά τέλος τελο προσθέμενη αξία που έχει αυτό το μέσο του Juncker για έργα υποδομών που ήδη είχαν χρηματοδότηση είτε μέσω επιχορηγήσεων είτε μέσω χρηματοδοτικών ε, μέσων τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν υπήρχαν μεγάλε διαφορέ δηλαδή. Η διαφορά που βλέπουμε εκ πρώτη όψεω είναι ότι οι επενδύσει που δεν θέλουν να κάνουν ε, τα κράτη-μέλη, δηλαδή να δώσουν χρήματα που δεν ξέρουν ακριβώς πού πηγαίνουν. Οι ακριβώ που προσφέρουν επενδύσει, συγκεκριμενα εργα ευρωπαϊκή προστέμενη αξία, που προσφερουν θέσει εργασία, αναπτυξη που εχουν μια σαφή κοινωνικο-οικονομική αξία και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, πολλαπλασιαστική δυνατότητα και σε πεδοτομέων και κλάδων, παραδείγματο χάρη, η ενεργειακή απόδοση, η βελτίωση του δικτύου μεταφορά κοινωνιών που γίνονται πιο καθαρέ είτε μέσω πλατών οδών, πλωτών οδών είτε μέσω σιδηροδρόμου Η βελτίωση των αστυνομικών κέντρων, η βελτίωση τη συνέργεια μεταξύ τομέων. Όλε αυτέ οι επενδύσει δεν πρέπει να πληγούν και να ε, υποστούν ε, αρνητικέ συνέπειε λόγω αυτού του επενδυτικού προγράμματο. Εμεί βλέπαμε ότι θα χρηματοδοτούνταν τέλο πάντων μετά τη ε, προθεσμία. Και ήδη από τον Ιούλιο μα είπε η Κομισιόν ότι χρηματοδοτούνται τα προγράμματα. Μα ανησυχεί λοιπόν αυτή η εξέλιξη. Εμεί θέλουμε η δική μα συνεισφορά να πηγαίνει σε έργα μεταφορών με ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, όπω είπα. Και το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και σε επίπεδο τομεακό να μπορεί να υπάρχει παρακολούθηση των έργων αυτών και των επένδυσεων από τις περιφερειακές αρχές. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Έχω ακόμη τέσσερις παρεμβάσεις. Θα τις ε, ακούσουμε εντός του χρόνου όμως. Ο κύριος Κωνσταφόρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και με τη σειρά μου εγώ θέλω να εξάρω τη σημαντική πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετά χρόνια αιμορραγεί από τον αποπληθωρισμό αλλά και από την μη έλευση της πολυποθούμενης ανάπτυξης. Προς αυτήν την κατεύθυνση δεν συνήργησε ούτε η Κομισιόν ούτε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τότε η σημερινή Επιτροπή ανταποκρίνεται κατά αυτόν τον τρόπο το χαιρετίζουμε. Όμω πρέπει να πούμε το εξή. Ακούεται πολύ καλά τα 315 δισεκατομμύρια και δημιουργούν ευθύνε και προσδοκίε. Οφείλω να σα πω ότι οι λαοί τη Ευρώπη είναι πολύ απογοητευμένοι το ότι η ανάπτυξη έμεινε σύστημα και δεν ήρθε ποτέ. Άρα είμαστε όλοι εντεταλμένοι σήμερα να καταστήσουμε επιτυχέ αυτό το εγχείρημα. Όμω για να μπορέσει να γίνει επιτυχέ αυτό το εγχείρημα των 315 δισεκατομμυρίων που φαντάζει ω έναν τεράστιο γίγαντα ανάπτυξη που όμω πρέπει να περπατήσει και να προχωρήσει και να μην καταρρεύσει, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Εγώ ακόμα μέχρι σήμερα δεν πήρα απαντήσει για ποια στοιχεία θα έχουμε όσον αφορά την ανάπτυξη συγκεκριμένων χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση πόσο θα μειωθεί η ανεργία. Τι έχουμε σήμερα, πρόβλημα ανάπτυξη και χάσμα ανάπτυξη γενικά και όριστα, ή έχουμε χάσμα ανάπτυξη μεταξύ βορρά και νότου. Ποιο είναι το πρόβλημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρε που έχουν ήδη ανάπτυξη να τι αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο και άκουσα και προηγουμένω ότι τα λεφτά πρέπει να πάνε στι χώρε εκείνε που έχουν πόρου. Άρα οι άλλε χώρε που μέχρι σήμερα δεν έχουν πόρου και μπήκαν σε μνημόνια να οδηγηθούν ουσιαστικά σε τριτοκοσμικέ χώρε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί τη δικιά μου χώρα Κύπρο θα μπορούσε με ένα δισεκατομμύριο μόνο ανάπτυξη, λεφτά η ανάπτυξη, αυτή τη στιγμή να ήταν έξω και από τα μνημόνια και να ήταν μια ευημερούσα χώρα. Πώ θα έρθουν αυτά τα λεφτά στη χώρα μου. Τελικά αυτά τα χρήματα θα πάνε αστόχευτα εκεί και όπου δεν υπάρχει πρόβλημα και να συνεχίζει να υπάρχει ακόμη αυτό το πρόβλημα της ανάπτυξης. Ένα άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να απαντηθεί. Θα μειωθεί η φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το πακέτο. Θα μειωθούν οι ανεργοί θα μειωθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει οι οποίε κλείνουν καθημερινά. Θα υπάρξει πραγματική ανάπτυξη στι χώρε εκείνε που δεν χρειάζονται. Θα υπάρξει μίκριση του χάσματο μεταξύ βορρά και νότου. Γιατί πιστεύω τελειώνοντα, κύριε Πρόεδρε ότι το χάσμα ανάπτυξη δεν είναι τα 315 δισεκατομμύρια αόριστα. Είναι το χάσμα ανάπτυξη που υπάρχει μεταξύ των χωρών, των βορείων χωρών και των νοτίων και για το οποίο μέχρι σήμερα δεν πήραμε καμία απάντηση μέσα από αυτό το πακέτο που ευελπιστώ πραγματικά να πετύχει. Ευχαριστώ. Σας είπα, για να λειτουργήσει το πρόγραμμα θα πρέπει και οι χώρες να εφαρμόζουν τις απαραίτητες ε, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Ο κύριος Δελανό, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ ε, ήμασταν ε, υπεράριθμοι αυτοί που θέλαμε ένα επενδυτικό πρόγραμμα για την Ευρώπη. Πολύ άριθμοι μάλλον. Αλλά διερωτώμεθα και έχουμε αρκετέ απορίε για το πρόγραμμα Juncker. Βεβαίω το καλό είναι ότι υπάρχει. Αλλά είναι μια πρωτότυπη εμπειρία, διότι ζητά το, από τον ιδιωτικό τομέα μια συμμετοχή με αναμενόμενο κέρδο βέβαια, αλλά και την εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια, ε, ένα πείραμα που καλό να το κάνουμε. Διότι μπορεί τελικά να έχουμε καλά αποτελέσματα και να βρεθεί η δυναμική όθηση που χρειάζεται η Ευρώπη με δημιουργία θέσεων απασχόληση. Εγώ όμω έχω τουλάχιστον δύο ερωτήσει από τι πολλέ απορίε μου. Πρώτα απ' όλα για το παράγοντα μόχλευση και τον πολλαπλασιασμό που αναμένουμε. Νομίζω ότι πράγματι πρέπει να βρούμε λύσει ώστε αυτό το στοιχείο, το πολλαπλασιαστικό, να, γίνει με παρεμβάσεις από το κράτος ίσως, από τις ε, τράπεζες, από κάποιες τράπεζες κρατικές ή από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάπως πρέπει να δικαιολογηθεί στα πλαίσια του παιδιτικού προγράμματος. Και δεύτερη απορία που δεν την έχουμε συζητήσει επαρκώς, αλλά πρέπει να την αναφέρω σήμερα, είναι η κατεπίγουσα ανάγκη. Χρειαζόμαστε κατεπηγόντως έργα, κατεπηγόντως οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση. Αυτό που εγώ όμως φοβούμαι είναι ότι τα έργα δεν θα είναι ακόμη ε, έτοιμα και ότι θα βρεθούν στις συμπληγάδες των ε, κρατών μελών. Δηλαδή, εδώ πρέπει να δούμε τι διοικητικά ζητήματα τίθενται ε, για τα κράτη-μέλη. Και τελευταία παρατήρηση. Δεν βλέπω πως ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την ανάπτυξη, για την έρευνα και την κοινοτομία μπορεί να συνδυαστεί με το επενδυτικό ε, πρόγραμμα Γιονκέρα. Ευχαριστούμε ο κύριος Πέτρης Ατάμα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι έχουμε ενώπιον μας μια τεράστια πρόκληση και θα έλεγα πως η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακυβεύεται εδώ. Δοκιμαζόμαστε αυτή τη στιγμή όχι μόνο από την οικονομία η οποία πάσχει, αλλά και από την επιστροφή της ε, γεωπολιτικής διάστασης με τη μορφή του Βλαντιμίρ Πούτιν και από την απειλή στην ίδια την ε, Ευρωζώνη, την πρόκληση μάλλον στην Ευρωζώνη. Το λοιπόν που επιχειρούμε να κάνουμε έχει τεράστια σημασία για το σύντομο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι χρήματα υπάρχουν για τις επενδύσεις και ότι υπάρχουν πακτολοί ιδιωτικού χρήματος που ψάχνουν που να πάνε και φυσικά έχει δίκιο. Τα κονδύλια υπάρχουν, όμως πιστεύω πως χρειάζεται να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να παρέμβουμε πολιτικά. Χρειάζεται να παρέχουμε το πλαίσιο, αλλά τίποτα παραπάνω. Καμία προτιμησιακή ε, μεταχείριση, καμία ε, κανένα περιθώριο λάθους. Πρέπει οι επενδύσεις να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν τους ε, επενδυτές σε αυτό και να δώσουμε αντικειμενικό, Τα διαφορετικά επενδυτές δεν θα έχουμε. Και θα ήθελα να πω στον ε, κύριο Έκχουτ ότι αν πραγματικά αυτό εννοείται όταν ε, είπατε να μείνουν έξω οι ιδεολογίες και οι ιδεολογικές αντιλήψεις, θα συμφωνήσω μαζί σας και να σας πω ότι και ο Μπιλ Κλίντον και ο Ντέιβιτ Κάρβερ, ο οποίος το είπε πρώτος, πραγματικά το θέμα είναι η οικονομία, βλάκα. Έτσι. Τελευταίος, ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα τρία σημεία. Το πρώτο αφορά το Μιγκέισον από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να εξασφαλίσουμε την επιχειρησιακή λειτουργία των προγραμμάτων το Connecting Europe Facility και το Ευρώπη 2020. γιατί τα πιο πολλά τους κονδύλια θα επαναναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν ε, για το, το Ταμείο Αγγίσεων του Ταμείου Στατικών Επενδύσεων. Τι λύση μπορεί να βρεθεί. Επαναχρησιμοποιούνται, χρησιμοποιούνται εκ νέου κάποια κονδύλια το Guarantee Instrument και το Risk Sharing Instrument της ε, ΕΤΕΠ. Γιατί μοιάζουν αυτά τα κονδύλια και αυτά τα, αυτοί οι μηχανισμοί. Επίσης θα πρέπει να, παραχθεί, να παραχθούν έσοδα για τον κοινωνικό προπολογισμό με αυτό το ταμείο και με αυτές τις επενδύσεις. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν στον κανονισμό διατάξεις συγκεκριμένε για το πώς τα κέρδη αυτά θα τροφοδοτούν τον ζωτικό προπολογισμό. Τρίτο σημείο. Δεξαμενή έργων, project pipeline. Φυσικά και πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Ούτε υπερρύθμιση ε, από τη μία, αλλά και σαφείς αρχές ε, και μέθοδοι λειτουργίας. Έχουμε πάνω από 2.000 έργα ε, που έχουν υποβληθεί. Τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν κάποια μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας ή μελέτη αντικτύπου που είναι σημαντικά στοιχεία για να μπορεί να συμμετάσχει ο δυτικός τομέας. Όπως είπε και ο Ότμαρ Κάρας, στηρίζω και εγώ στο ότι θα πρέπει να μην υπάρξει καμία πολιτική εμπλοκή, πολιτική συμμετοχή. Αν θέλουμε να είναι ελκυστικά τα project για τον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να υπάρχουν επίσης διαφανή κριτήρια για την επιλογή αυτών των έργων και θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ τομεακής διάστασης να εκπληρώνουν τα έργα, δηλαδή ε, τους στόχους του Connecting Europe και του 2020 και να έχουμε οικονομική ε, μελέτη, μελέτη οικονομικού αντικτύπου. Στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης, να μην έχουμε μόνο συγκεκριμένα για πόσα χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομο παραδείγματος σε μια περιοχή, αλλά αντίκτυπο, μελέτη αντικτύπου, για να ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα έχουν αυτά τα σχέδια στα οποία επενδύουμε. Ευχαριστώ. Λέω πρόεδρο, ολοκληρώνουμε εδώ αυτή την συνεδρίαση. Τέθησαν πολλά ζητήματα. Ε, θα τα προσθέσουμε στα 110 ερωτήματα τα οποία προέρχονται από τις περισσότερες εξημών και τα οποία έχουμε διαβάσει. Έχουν διαβαστεί σε επιτροπές. Θα σας απαντήσουμε μέσα στις επόμενες ώρες. Να πω ότι έχουμε και μία συνάντηση ερωταπαντήσεων στις 26 Φεβρουαρίου από τις 2 τις 4. Την επόμενη Πέμπτη λοιπόν θα είναι παρόντες οι εκπρόσωποι εμπειρογνώμονες ε, της Επιτροπής που θα απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα. Θέλω να ευχαριστήσω και την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, που έχουν εκπροσώπους τους εδώ σήμερα και να δώσω τώρα το λόγο στους δύο συνεισηγητές για να μας πούν πώς ε, είδαν αυτή την ανταλλαγή απόψεων και ποια κατεύθυνση θέλουν να δώσουν στις εργασίες μας. Να δώσω ανάποδα πλέον το, το πρώτο στον κύριο Φερνάντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους. Σημειώνουμε τα σχόλια και θα τα λάβουμε σοβαρός υπόψη. Αλλά αυτό που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε είναι ότι το πρόγραμμα Juncker, το Ευρωπαϊκό Αυτοταμείο Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ, για το οποίο συζητάμε, είναι ότι θα πετύχει, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Και κανείς δεν μπορεί να πει ότι θα αποτύχει κιόλα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι απλώς ότι θα κερδίσουμε σίγουρα, εάν λάβει σάρκα και ωστά θα κερδίσουμε με μία συμβολή 800 εκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Τουλάχιστον έτσι θα έχουμε μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων και κινητοποίησή τους και έτσι θα έχουμε αυτήν την ε, προσφορά κινήτρων που θέλουμε. Αυτά τα 8, τα τα 8 δις ευρώ που θα προβλέψουμε θα είναι η σκανδάλι που θα κάνει το όπλο να εκπυρσοκροτήσει και να κινητοποιηθούν πλέον οι επενδύσεις. Ε, θα έχουμε με το πρόγραμμα αυτό ανάπτυξη, απασχόληση, μια Ευρώπη ισχυρότερη, μια Ευρώπη πιο αλληλέγγυα. Ακούστηκαν αρκετές ε, επικρίσεις φαντάζομαι ότι θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μόχλευση. Τα έχει πει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο παράγοντας μόχλευσης 15 θα, ε, είναι κάτι που θα προκύψει εξ ορισμού διότι ως τώρα με τα άλλα προγράμματα, με το κόσμο, λόγου χάρη ή άλλα, με παράγοντα πολλαπλασιαστικό 28, είναι στοιχεία που μπορούν να απαντηθούν με τεχνική τεχνικές, ε, με τεχνικούς υπολογισμού. Το έχει δείξει η εμπειρία μας από το πρόσφατο παρελθόν. Προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν ήταν διαφορετικά από αυτό που συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπούλμαν. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σα θυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περίμενε πάρα πολύ καιρό μια τέτοια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις ε, εκθέσεις της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας, ιδιαίτερα στην έκθεση των συναδέλφων Κάρας και Τάισεν, ο οποίος σήμερα είναι μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε ζητηθεί από την ε, Κομισιόν να αναλάβει ε, περισσότερο προορατικό ρόλο στην δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων απασχόλησης και βιώσιμης ανάπτυξης. Και τώρα πραγματικά το έχει κάνει πραγματικότητα και πολύ καλώς έπραξε είδα μια ειλικρινή δέσμευση από όλες τις πλευρές για να δημιουργηθεί κάτι καλό και πραγματικά ε, παρότι υπήρξαν έτσι κάποιες ε, μικρές ε, εχμές για ιδεολογίες, πολιτικές και τα λοιπά, πιστεύω πως όλοι έχουμε την επιθυμία να δημιουργήσουμε ένα πολύ καλό προϊόν, ένα καλό αποτέλεσμα και γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσω να εργαστώ όσο το δυνατόν πιο σκληρά τις επόμενε εβδομάδες και μήνες. Ευχαριστούμε. Μπορούμε να κηρύξουμε τη λήξη αυτής της πρώτης ε, συνεδρίασης. Να διευκρινίσω ότι το επόμενο ραντεβού μα είναι την Δευτέρα 2 Μαρτίου από τις 3.30 και μισή έως τις 6.30 για μια σειρά από ακροάσεις. Και έπειτα την παρουσίαση του σχεδίου ε, έκθεσης ε, στις 12 Μαρτίου στο Στρασβούργο. Ρομπερτό, ε, νομίζω ότι θα κλείσουμε με αυτά και καλώ τους συντονιστέ της Επιτροπής Προπολογισμών να παραμείνουν σε αυτή την αίθουσα.